So then we start uh, the meeting. The first item is adoption of the uh, agenda. I have uh, no... Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Can we adopt it as is? Yes, thank you. Πρώτο θέμα έγκριση της ημέρησιας διάταξης. Δεν έχουμε καμία πρόταση τροποποίησης. Εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη βδομάδα και την επόμενη έχουμε τις ακροάσεις των νέων επιτρόπων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δύο αποτελούν βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΝΤΕΒΕ. Είναι όλες οι ακροάσεις δημόσιες και θα μεταδοθούν και στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να σα πω λίγα λόγια για τη διαδικασία. Στην CCC, ε, διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών, είχαμε σχετική συζήτηση ε, για το σε ποια επιτροπή θα είναι αρμόδια, ποια θα είναι προσκεκλημένη, ποια θα είναι συνδεδεμένη κλπ. Στην ακρόαση του κάθε επιτρόπου. Κάθε επιτροπή θέλει φυσικά να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Είχαμε λοιπόν μια διαδικασία ε, σύμφωνα με την οποία έχουμε τη βασική αρμοδιότητα για δύο επιτρόπους. και είμαστε προσκεκλημένοι και σε άλλε επιτροπέ. Θα σα περι... σας ε, τα αναφέρω αυτά τώρα και μετά θα σα μιλήσω για τη διαδικασία. Οι δύο βασικέ ακροάσεις που θα έχουμε θα είναι με την κυρία Γιούτα Λάινεν, ε, επίτροπο για την Διεθνή Συνεργασία, αύριο από τι 9 έω τι 12. Και να επαναλάβω, 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ακόμα και αν δεν είναι κανείς παρόν, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, διότι θα είναι αδύνατον, σας διαβεβαιώ, θα είναι αδύνατον για τους ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις εάν δεν ξεκινήσουμε στις 9. Θα πρέπει συνέχεια να χτυπάω το σφυράκι για να ε, περιοριστείτε στον χρόνο ομιλία σας. Να το ξέρετε λοιπόν αυτό. Και θα προσκληθούν οι εξή επιτροπές να συμμετάσχουν η ΑΦΕΤ, η ΙΝΤΑ, η ΛΥΜΠΕ και η ΦΕΜ. Είχαμε συζήτηση, είπαμε ότι θέλουμε επιπλέον χρόνο, θα έχουν χρόνο ομιλίας, ε, αυτό δεν ήταν δυνατό, γι' αυτό εναπόκειται στις ε, πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν αν θα τους δοθεί ε, χρόνος ομιλίας και αυτό ισχύει σε όλες τις επιτροπές. Στις περισσότερες επιτροπές, η προσκεκλημένη επιτροπή δεν θα έχει χρόνο ομιλίας. Αλλά στην ΤΕΒΕ μπορεί να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό εναπόκειται στι πολιτικέ ομάδε να το αποφασίσουν. Επίση, θα έχουμε ακρόαση του κυρίου Γιάννη Λενάρτση ε, για τη διαχείριση των κρίσεων. Ε, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου από τις 6.30 έως τις 9.30. Η Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι συνδεδεμένη επιτροπή στην ακρόαση αυτή. Εμεί δε είμαστε προσκεκλημένοι στις εξή ε, ακροάσει, ε, του Φιλ Χόγκαν, ε, νέου Επιτρόπου για το Εμπόριο, σήμερα στι 6.30 με 9.30 του Βιρτζίνιους Σινκεβίτσιους, νέου Επιτρόπου για το Περιβάλλον και τους Οκεανούς, την 5η από τις 2.30 έως τις 5.30 και του Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπροέδρου για Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, 5η από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 και του Γιώζεπ Πορέλ, ε, αντιπροέδρου και ε, νέου ε, είπα του εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Δευτέρα 7 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 5.30. Επίσης έχω μια ανακοίνωση για το βραβείο Ζαχάροφ. Συνάδελφοι, παρακαλώ να θυμάστε ότι σήμερα στις 5 η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ θα έχει μια κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ και την ΤΡΟΑ για παρουσίαση των υποψηφιωτήτων για το βραβείο Ζαχάροφ θα μεταφερθούμε σε άλλη αίθουσα, στην PHS 3C50. Δεν γνωρίζω που είναι, λέει ο πρόεδρο. Ε, νομίζω όμω ότι ε, θα σα ε, βοηθήσουν κάποιοι να βρείτε το δρόμο. Επίση, θα έχουμε κοινή ψηφοφορία, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, για τι υποψηφιότητε στι 8 Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αποφασίσετε τίποτα σήμερα. Και τέλος, να σας πω ότι έχουμε κοινή ψηφοφορία για την πιθανή έναξη τριμερούς διαλόγου για το ε, ε, ε, εργαλείο για την γειτονία, την ανάπτυξη και την διεθνή συνεργασία στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί. Είναι καθαρά τεχνική σε φύση η ψηφοφορία και θα πραγματοποιηθεί πριν την ψηφοφορία για το βραφείο Ζαχάροφ. Θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες ε, εν ευθέτω χρόνο. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 3, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Ωραία, προχωράμε. Στο σημείο 4. Οι πολιτικέ ανθρωπιστική βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν κόσμο με ε, περισσότερε ανάγκε και περιορισμένου πόρου. Είναι μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Ξέρω ότι οι σχέσεις ε, της Επιτροπής ΔΕΒΕ με τον Επίτροπο έχουν λειτουργήσει εξαιρετικά καλά τα τελευταία πέντε χρόνια. Εγώ βέβαια είμαι νέος πρόεδρος, αλλά το πιστεύω. Είναι μεγάλο προνόμιο να σας έχουμε εδώ μαζί μας ε, σήμερα για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Τελευταία φορά που ήρθατε στην Επιτροπή μας, ε, κύριε Επίτροπε, τον Φεβρουάριο, ήταν ε, σε μια ε, ε, δημόσια κρόαση για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θέλουμε άλλη μια γενική συζήτηση, ώστε τα νέα μέλη της Επιτροπής μας να έχουν μια εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 130 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανάγκη από βοήθεια και οι ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο και ε, παρέχει περισσότερο από το 1,5% ε, που, που ζητάνε το Ηνωμένα Έθνη σε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό βέβαια μας κάνει υπερήφανους, είναι όμως και σημαντική ευθύνη για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να παρακολουθούμε την σωστή χρήση των πόρων αυτών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να μας ε, παρουσιάσει τα όσα ε, έχουν πραγματοποιηθεί κατά διάρκεια της θητείας του, να μας περιγράψει τις προκλήσεις που μας περιμένουν και κατόπιν θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Thank you so much, ε, Chair. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Συναντηθήκαμε και στην Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα στην ΟΚΑ Και πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ε, επικοδομητική αυτή η σύντομη περίοδος των ε, συναντήσεων. Είδαμε λοιπόν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πώς διαμορφώθηκαν στην πράξη σε ένα πολύ απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Και πιστεύω ήσασταν και εσείς παρόντες στην ΟΥΝΚΑ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ λοιπόν, σημαντική η παρουσία μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εικόνα μας Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, γιατί θυμάμαι πριν από πέντε χρόνια Ο βουλευτή. Και φυσικά χαίρομαι που βλέπω και κάποιους ε, παλιούς καλούς φίλους, Κύριε Σνόερ, για παράδειγμα, Και βλέπω επίση πολλού νέου συναδέλφου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συναντιόμαστε για να υπάρξει μια υπέρβαση των συνηθισμένων πρακτικών, γιατί έτσι έχει η πολιτική ζωή και έτσι έχει κυρίως ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Πριν από πέντε χρόνια λοιπόν, ακριβώς πέντε χρόνια μάλιστα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 για πρώτη φορά εμφανίστηκα ενώπιον της Επιτροπής σας. Επρόκειται τότε για την ακρόαση για την επιβεβαίωση της ανάλυσης των καθηκόντων μου. Ήταν λοιπόν, αν θέλετε, η σημερινή ημέρα μια επέτειος. Εκείνη την ημέρα λοιπόν συνειδητοποίησα και αντιληφθήκα πόσο σημαντική και από τη δική μου εμπειρία ως υπουργό, ως ε, εθνικός βουλευτής, ως ευρωβουλευτές. Κατανόησα λοιπόν πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή αυτή. Γιατί η δουλειά σας και η δουλειά μας ξεπερνά κατά πολύ την πολιτική και τις αποφάσεις για χρηματοδότηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή ΔΕΒΕ θεωρώ ότι αποτυπώνει τις πιο ευγενείς αξίες της Ένωσης μας και όπως τόνισε επανελειμμένα ο Ζαν Κλοντία το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το να δίνουμε στους ε, πλέον ε, αδύναμους ε, μία ευκαιρία και αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από την εθνότητά τους, από την σκία τους από την σεξουαλική τους ε, ταυτότητα. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε αυτή την ε, μεγάλη πολιτική οικογένεια και πραγματικά είμαι υπέρμαχος ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας της οικογένειας αυτής και είμαι βέβαιος ότι θα απολαύσετε τη σύνδεση αυτή, τις επαφές αυτές με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τόσο μεγάλη δέσμευση για τις κοινέ μας αρχές και τις κοινέ μας αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγαπητοί φίλοι. Όλοι γνωρίζετε ότι τα ανθρωπιστικά μέσα δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Αλλά να πούμε ότι αυτά τα πέντε χρόνια, χάρη στην υποστήριξή σας, χάρη στην υποστήριξη της Επιτροπής σας, ε, δεν πρέπει να τρεπόμαστε να το τονίσουμε, και χάρη και στην ε, αγαπητή γραμματεία, καταφέραμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου. Και αυτό σήμαινε ότι μπορέσουμε να ανακουφίσουμε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να εστιαστώ σε τρεις ε, περιπτώσεις, σε τρία συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν θέλετε το κλειδοδότημά μου ή το κοινό μας κλειδοδότημα, αγαπητοί φίλοι. Τρία λοιπόν κρίσιμα παραδείγματα. Η κρίση έμπολα στην Δυτική Αφρική πριν από πέντε χρόνια. Κατάρτιση σε κατεπίγουσες καταστάσεις και τρίτον το Rescue που από κοινού καταφέραμε να αναβαθμίσουμε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας ξεκινήσουμε με την κρίση έμπολα στη Αφρική και φυσικά να φωτίσουμε και κάποιες άλλες πτυχές της κρίσης αυτής. Η κρίση αυτή αποτέλεσε ένα ορόσημο εκατοντάδες άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους σε καθημερινή βάση. Άλλαξε η όλη κρίση τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις ε, κατεπίγουσες ε, καταστάσεις σε ό,τι αφορά την υγεία και το πώς αντιδρούμε σε αυτές κυρίως. Η πρώτη μου λοιπόν δέσμευση προς το Κοινοβούλιο εδώ την ίδια ημέρα, πριν από πέντε χρόνια ακριβώς, ήταν να πάω και να επισκεφτώ τις τρεις χώρες που πλήχθησαν από την κρίση έμπολα, Λιβερία, Σιερελεώνα και Γουινέα. Και θυμάμαι την πρώτη ακρόαση, την πρώτη μάλλον συνεδρίασή μου εδώ ήταν για το έμπολα. Μου τρέφησε λοιπόν το ερώτημα από έναν Κροάτη, αν δεν κάνω λάθος, και με ρώτησαν λοιπόν ποια θα ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στα πλαίσια της κρίσης έμπολα. Απάντησα κατευθείαν ότι ναι, θα πάω να επισκεφθώ τις χώρες αυτές, θα παρευρεθώ επί τόπου για να μπορέσω να αξιολογήσω την κατάσταση. Και ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, να σας πω ότι η απόφαση αυτή ήταν ε, πολύ καλή. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο κρίσιμες ε, καταστάσεις από τα γραφεία μας στις Βρυξέλλες. Η κρίση λοιπόν έμπολα στη Βετική Αφρική αποτέλεσε μια δοκιμασία για τη διεθνή κοινότητα και μας δίταξε ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε καταστάσεις και κρίσεις όπως ο έμπολα. Κινητοποίησαμε και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και οικοδομήσαμε ε, μια εγκατάσταση ε, ιατρικής ε, εκένωσης ε, που ήταν καθοριστικός παράγοντας για να πείσουμε πιο πολλοί ε, γιατρούς και ιατρικό προσωπικό να παρευρεθούν εκεί. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η πολιτική πρωτοβουλία. Ήταν λοιπόν ένα από τα κρίσιμα κενά χάσματα τα οποία εντόπισα κατά την επίσκεψή μου και γι' αυτό επιμένω ότι χρειάστηκε να επισκεφτώ τις χώρες αυτές γιατί μόνο τότε συνειδητοποιήσαμε ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνηση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό επί τόπου. Και ασφαλώς μάθαμε και τα μαθήματά μας. Καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ιδρικέ ομάδε έτοιμε, να αναπτυχθούν ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα για τέτοιες κατεπίγουσες ε, περιπτώσει. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το Ιατρικό Σώμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ, για να είμαι δίκαιος, προς δύο εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, τον, προ, τον τρέχοντα πρόεδρο της Γερμανίας Στάινμαρ ε, και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς, ο οποίος με υποστήριξε τόσο πολύ στην δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος. Πλέον λοιπόν το σώμα αυτό αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και αποτελεί την άμεση αντίδρασή μας για τέτοιες προκλήσει που χρειάζονται άμεσα κινητοποίηση ιατρικού προσωπικού όταν ιδιαίτερα οι εθνικές, οι εθνικοί πόροι έχουν ε, εξαντληθεί. Ε, το Ευρωπαϊκό λοιπόν Ιατρικό Σώμα ενισχύει την ε, δυνατότητα αντίδραση, κατεπίγουσα αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το αποδείξαμε επί τόπου. Κοιτάξτε το παράδειγμα, για παράδειγμα, τη του ξεσπάσματος του ιού έμπολα το 2018 στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό. Το 2018 καταφέραμε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού σε τρεις μήνες. Και αν ε, συγκρίνουμε το τι έγινε με πριν από πέντε χρόνια, πραγματικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Φυσικά, κάθε φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και τώρα αντιμετωπίζουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη, τα δεύτερα μεγαλύτερα κρούσματα έμπολα στην ιστορία και τα πράγματα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά γιατί φυσικά είναι μία μάχη κατά του χρόνου αλλά υπάρχει και μία χρόνια αστάθεια η οποία επικρατεί και αυτό προφανώς και δυσκολεύει περαιτέρω την δουλειά μας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εμπόδια σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, πολλοί περιορισμοί και φυσικά χρειαζόμαστε πιο αμα, προσαρμοσμένες ε, λύσεις και παράλληλα χρειαζόμαστε και πιο πολύ χρόνο προφανώς. Έχουμε όμως επιτόπου πιο πολύ προσωπικό. Έχουμε πιο αποτελεσματικά εμβόλια που έχουν ε, αποτελεσματικές ε, λύσεις αποτελούν μια αποτελεσματική λύση και γενικά υπάρχει πιο πολύ υποστήριξη σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Είναι λοιπόν μεγάλε οι διαφορές και προφανώ, εδώ μπορώ να το αναφέρω αυτό, η κατάσταση είναι καλύτερη σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματικότητα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Τότε, το πιο σημαντικό διεθνές ε, εργαλείο. Ο διεθνής πυλώνας αντιμετώπιση τέτοιων ιατρικών κατεπούσεων καταστάσεων ήταν σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση τότε, πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, πλέον, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Είναι πιο αποτελεσματικά και γι' αυτό από την αρχή της νέας θητείας του Δ. Τέτρους υποστηρίξαμε τις προσπάθειές του για την ατζέντα μεταρρύθμισης της ΠΟΗ. Δεύτερη πρόκληση και παράλληλα δεύτερη κατάκτηση σε ό,τι αφορά την κατάρτιση σε κατεπίγουσες περιπτώσεις. Οι συνάδελφοί μου επιμένουν ότι έχω παθιαστεί με καλό τρόπο με το θέμα αυτό. Το δέχομαι αυτό ως ε, αξιολόγηση, γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάποιες θετικές ε, τέτοιες ε, στη ζωή μας. Πώς να το κάνουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελεί το πιο θεμελιώδες στοιχείο της ζωής μας. Αυτό με βρίσκει απόλυτα πεπισμένο. Μία μέση ανθρωπιστική κρίση κρατά πάνω από εννέα χρόνια. Τέτοιες καταστάσεις παρατεταμένης έκτακτης ανάγκης δεν αποτελούν πλέον την εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Πάνω από 65 εκατομμύρια παιδιά πλήττονται σε τέτοιες καταστάσεις ε, έκτακτης ανάγκης. Τα παιδιά αυτά δεν εκπαιδεύονται. Δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν προστασία και δεν έχουν κάποια ελπίδα, κάποια προοπτική για το μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν τα διαπίστωσα επανειλημμένα σε όλους μου τις επισκέψεις επί τότου και έχω πολλές α, ε, τέτοιες ε, αναμνήσεις οι οποίες με θλίβουν ιδιαίτερα στην Συρία, στο Ιράκ, στο Σαχέλ διαπιστώνω ότι η εκπαίδευση δεν ε, αποτελεί μόνο μία ανάγκη μεσοπρόθεσμη, αποτελεί μία ανάγκη για την ε, επιβίωση των ανθρώπων. Το 2015, λοιπόν, μόνο 1% της ανθρωπιστικής μας βοήθειας κατευθυνόταν ε, στην εκπαίδευση. Κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Τότε λοιπόν ε, έκανα μία ε, υπόσχεση να αυξηθεί η υποστήριξή μας αυτής και για να δημιουργηθεί μία ασπίδα, μία ασπίδα κατά της βίας, μία ασπίδα κατά της καταναγκαστικής εργασίας, κατά των ε, καταναγκαστικών γάμων και φυσικά κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Πετύχαμε αποτελέσματα. Φέτος, 10% της ε, αρρωγής μας απευθύνεται σε θέματα εκπαίδευση σε τέτοιε καταστάσει εκτακτού ανάγκη. Πάνω από 165 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για παγκόσμια ρεκόρ σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση σε τέτοιε καταστάσει εκτακτού ανάγκη. Από το 2015 και 2019 επενδύσαμε πάνω από 450 εκατομμύρια σε εκπαίδευση σε τέτοιε καταστάσει εκτακτού ανάγκη. Πιάσαμε τα 6,5 εκατομμύρια παιδιά σε 55 χώρες. Και μιλώ στο πρώτο πληθυντικό. Εμείς. Και επιμένω σε αυτό το εμείς, γιατί ήταν η Επιτροπή σας αυτή που ζήτησε πιο πολύ δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό για να υπάρξουν πιο πολλοί πόροι χρηματοδότησης για εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτακτού ανάγκης. ask us to do something else, to come forward with... Δηλαδή, ε, να ξεκινήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με την εκπαίδευση σε αυτές τις ε, επίγουσες καταστάσεις και εμείς το κάναμε. Τον Μάιο του 2018 εγκρίναμε την πρώτη ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτού του είδους την εκπαίδευση που, μας, που καθοδηγεί όλα τα προγράμματά μας, τα προγράμματά μας επιτόπου και όλες τις εταιρικές μας σχέσεις έτσι ώστε να υπάρχει ένας ευέλικτος και συντονισμένος τρόπος λειτουργίας ε, επιτόπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε ένα υψηλό επίπεδο ε, χρηματοδότησης. Η δέσμευσή μας είναι να ξαναφέρουμε τα παιδιά στο σχολείο μέσα σε τρεις μήνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς βρήκαμε αυτό το συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο μετά από ε, πολλές και μέσα από πολλές επιστημονικές αναλύσεις. Μπορώ να συνεχίσω. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την μετάφραση. Όλα καλά τώρα. Πολύ ωραία. Μπορώ να συνεχίσω λοιπόν. Έχω πει επανειλημμένα ότι θα πρέπει ε, να μην επιτρέψουμε να χαθεί οποιαδήποτε γενιά. Αυτή, ε, αυτό είναι το, το, ο στόχος μας και αυτός, ε, αυτή είναι η ηθική μας υποχρέωση. Τρίτο σημείο και τελευταίο παράδειγμα σχετικά με την εξαιρετική συνεργασία μας με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ είναι το Rescue αυτό δηλαδή το αναβαθμισμένο σύστημα, ο αναβαθμισμένος μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική προστασία ανθρωπιστικές ε, ε, κρίσεις ε, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα βίας και πολέμου. Μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών που είναι όλο και πιο περίπλοκες, όλο και πιο έντονες και δύνατον να προβλεφθούν. Και ναι, αυτό συμβαίνει λόγω της κλιματικής αλλαγής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι fake news. Όχι, καθόλου fake news δεν είναι. Ζούμε κάθε μέρα τον αντίκτυπο της ε, και την επίδραση της, της κλιματικής αλλαγής παντού, κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, ε, η δικιά μου θέση ως Επιτρόπου έχουμε ένα στόχο, να βοηθήσουμε να σωθούν ζωές επιτόπου και να δείξουμε στους πολίτες μας, στους δικούς μας αλλά και τους πολίτες όλου του κόσμου ότι δεν αφήνουμε κανέναν στην τύχη του μετά από μια καταστροφή. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2017 μια μακροσκελή διαδικασία μετά από μια πολύ κακή ε, εμπειρία στην Πορτογαλία, θα τη θυμάστε φαντάζομαι όλοι, αποφασίσαμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας ε, στην Ευρώπη με τη δημιουργία του RESC EU ε, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έναν, ε, ένα δίχτυ προστασίας για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη διάρκεια κρίσεων. Το προηγούμενο Μάρτιο, έξι μήνες πριν, λήφθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί και μία μεταβατική ένα αέρια, ένας ε, αέριος στόλος ε, για την καταπολέμηση των δαστικών ε, πυρκαγιών και βοηθήσαμε με Καναντέρ της Ιταλίας και της Ισπανίας και με τον τρόπο αυτό σώσαμε ζωές στην Ελλάδα πριν από δύο μήνες και βεβαίως αυτή ήταν η πραγματική ε, αλληλεγγύη, την οποία είδαμε και την εκφράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλβανία, αλλά και στη Βολιβία ακόμα, μετά από τις ε, σοβαρές πυρκαγιές ε, στον Αμαζόνιο. Και φυσικά το καλοκαίρι του 18 στην χώρα σας, στη Σουηδία, γιατί και τότε ήμουν παρόν. Πριν από την πραγματική αναβάθμιση του Rescue και πριν δημιουργηθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά και στην Σουηδία το 2018 συνειδητοποιήσαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι κάτι απτό και συγκεκριμένο. Και να σας πω και ένα ανέκδοτο, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην ε, Κύπρο συνάντησα Σουηδούς που με αναγνώρισαν ε, από τις ε, συνεντεύξεις που είχα δώσει στην <laughs> τηλεόραση της Σουηδίας ε, και μου λέγανε «Α, Επίτροπε, είσαι ο ήρωάς μας, γιατί ε, βοήθησε στη χώρα μας. Αυτό είναι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Ε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρνει να δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή που αυτή η βοήθεια είναι απαραίτητη. Το κάναμε λοιπόν ε, σχεδόν δύο χρόνια πριν στην, και στην χώρα σας. Επομένως αυτός ο νέος μηχανισμός προστασίας, πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και βεβαίως Τώρα συζητούμε ε, και το μέλλον του RESC EU ε, και νομίζω ότι αυτή πλέον είναι η δικιά σας ε, αρμοδιότητα να ξεπεράσετε τα όσα έγιναν μέχρι τώρα. Να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιατρικές κρίσεις όπως αυτό της έμπολα αλλά βεβαίως και οποιαδήποτε, οποιαδήποτε ατυχήματα BRN. Οποιαδήποτε προκύψουν το Τσερνόμπιλ δεν είναι και τόσο παλιό όσο πιστεύουμε. Επομένως, χρειαζόμαστε κοινή ε, ε, ευρωπαϊκή αντίδραση. Ε, ακόμα τη χρειάζονται και οι μεγάλες και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα πρέπει να είμαστε μαζί γιατί η καιροί είναι δύσκολη. Και βεβαίως δεν συζητούμε μονάχα για την αποτελεσματικότητα αλλά και την οικονομία κλίμακας θα είναι πιο φτηνό για όλους μας και πιο συμφέρον για όλους μας. Επομένως, το Rescue είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο, το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, πολιτικής ε, προστασίας ε, και χαίρομαι που έχουμε συμπεριλάβει και αυτό στις επιτυχίες της Επιτροπής Juncker και αυτό οφείλεται οπωσδήποτε και στην πολλαπλή συνεργασία μας ε, με την επιδίωξη κοινών στόχων. Και θυμάμαι ότι άκουσα πολλές ε, συμβουλές από, συναδέλφους εδώ και από γερμανούς συναδέλφους που μας έλεγαν ότι έπρεπε ε, να επισκεφθούμε όλα τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας έτσι ώστε να πείσουμε ε, τα τοπικά κοινοβούλια, τα ομοσπονδιακά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις έτσι ώστε να δώσουν το πράσινο φως όλοι. Μαζί λοιπόν επιτύχαμε αυτόν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο και ένας από τους καλούς μου φίλους ε, στην Κομισιόν, από τους συναδέλφους μου είπε ότι πραγματικά ξεπεράστηκε οποιαδήποτε προσδοκία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτά που σας ε, ανέφερα ήταν τρία συγκεκριμένα παραδείγματα από προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά επιτόπου. Δυστυχώς όμως οι κρίσεις είναι πολλαπλές. Υπάρχουν 132 ε, εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστική αρρωγή το 2019 οι εκτοπισμένοι έχουν φτάσει στα 69 εκατομμύρια και αυτό είναι ένας αριθμός χωρίς προηγούμενο. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που βρέθηκε πραγματικά στην πρώτη γραμμή ανταπόκρισης ε, ε, της ανθρωπιστικής κρίσης στην Συρία με 17 δις βοήθεια τα τελευταία 8 ε, χρόνια. Στην ΟΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε για μία ακόμα φορά να κάνουμε την διάσκεψη για την Συρία και αποδείξαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη, στρατευμένη στην επίλυση αυτής της κρίσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που ηγήθηκε της διεθνούς υποστήριξης στις χώρες της περιφέρειας, της περιοχής αυτής, ε, όπως η Τουρκία, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ιράκ και η Αίγυπτος, που υποδέχτηκαν 6 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Συρία και αλλού. Ήταν ε, μία από τις δικές μας επιτυχίες ε, ε, επίσης αυτή η εφαρμογή της πολιτικής μας μέσω της διευκόλυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δύσκολη η κατάσταση, ωστόσο καταφέραμε να ανακουφίσουμε τον πόνο των ανθρώπων στην Τουρκία τα τρία τελευταία χρόνια με πολύ ικανοποιητικό, επιτυχημένο τρόπο και φυσικά καταφέραμε ε, να συνδέσουμε και την ε, εκπαίδευση με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο ε, σκέψης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπρέπεια των προσφύγων, αλλά και πολύ σημαντικό και για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρουμε δηλαδή να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας, τις διαφωνίες μας όσον αφορά το resettlement και το relocation. Μπορώ επίσης να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία για πρώτη φορά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 2016 ε, έδωσε και ε, ε, βοήθεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στους ετούντες άσυλο στην Ελλάδα και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αλλά και ας μην λησμονούμε ότι πάλι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που ήταν παρούσα ε, στο πλευρό των πιο ευάλωτων ε, και πιο λησμονημένων. Αναφέρομαι στις λιουσμονισμένες ε, ε, κρίσεις που αποτελούν σημαντική πρόκληση ε, για, για σας στην επόμενη θητεία σας. Και μπορώ να πω μέσα από την εμπειρία μου ότι θα πρέπει να επιμείνετε πολύ σε αυτήν την πολιτική έτσι ώστε να δίνετε βοήθεια στις λισμονημένες κρίσεις. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν συνδιοργανωτής της πρώτης διάσκεψης για την ε, ε, δημοκρατία του Κονγκό την προηγούμενη την προηγούμενη χρονιά και κατάφερε να μαζέψει χρήματα έτσι ώστε ας πούμε να υλοποιηθούν προγράμματα όπως είναι το νοσοκομείο Πάντζη το οποίο λειτουργεί ο Δόκτωρ Ντένις Μουκβέγγε Νόμπελ ε, ειρήνης. Επίσης, την, τελευταία, την προηγούμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία ασχολήθηκε με τους Ροχίνγκα στην ε, Μιανμάρ. Και ήμουν ο πρώτος ε, υψηλού επίπεδου πολιτικός που επισκέφθηκα το Rakhine State τον Μάιο του 2017 πριν από την μαζική έξοδο των 700.000 Ροχίνγκα από εκεί προς τον Μπαγκλαντές που έγινε μετά από τρία μήνες. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία αποτέλεσε, ε, ήταν ο συνδιοργανωτής της διάσκεψης για τους Ροχίνγκα, ε, όπου μαζεύτηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει μέσα από αμεροληψία, από ανεξαρτησία, αλλά οπωσδήποτε με ανθρωπιά να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Αγαπητοί φίλοι, οι ραγδαία αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες και οι περιορισμένοι πόροι μας ε, μας έχουν κάνει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που προσφέρουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Στην τελευταία συνάντηση με τους προκατόχους σας, είπα ότι το πώς παρέχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια είναι συχνά εξίσου σημαντικό με τη βοήθεια αυτή καθ' αυτή. Ναι, πράγματι πρόκειται για πρώτες βοήθειες και σα το λέω αυτό ο γιατρός. Ε, είναι παρόμοια η κατάσταση και επέμενα να έχουμε πιο καινοτόμα ανθρωπιστική βοήθεια, πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη. Το ίδιο σας λέω και σήμερα. διότι με τις αρμοδιότητές σας ως μέλη ε, του, του Κοινοβουλίου θα αντιμετωπίσετε πολλές σημαντικές προκλήσεις ε, στο εγγύς μέλλον και σημαντικά θα πρέπει να αποφασίζετε πάνω σε επίμαχα θέματα. Έχετε όμως τη σοφία, την εμπειρία και τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης για να λάβετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις σε κάθε, σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποια από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να παρέχουμε πιο καινοτόμε, πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την βοήθεια σε μετρητά, που είναι εξαιρετική η απάντηση στην ερώτηση αυτή. Ε, είναι ο ορισμός της ε, ε, γρήγορης, άμεσης και ευέλικτης βοήθειας. Επιτρέπει στους ανθρώπους να καλύψουν ε, τις καθημερινές τους ανάγκες ε, αυτόνομα και με αξιοπρέπεια. Έχουμε αλλάξει λοιπόν ε, τον τρόπο παροχής της βοήθειας από το 10% 100 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 2011 σε σχεδόν 40% 900 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και το ίδιο κάνουμε και το 2019 έχει λειτουργήσει στην Τουρκία, στο, στη Ιορδανία, τη Σομαλία, την Ουγγάντα και την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει καλά και αλλού. Νομίζω ότι ήδη μακρηγόρησα. Ήθελα όμως ε, να σας παρουσιάσω τις προσωπικές μου εμπειρίες ε, κατά τη διάρκεια της ε, θητείας μου και να σας μεταφέρω κάποιες σημαντικές ε, παρατηρήσεις μου και νομίζω ότι αυτά θα είναι χρήσιμα και για σας. στο δύσκολο χρονικό διάστημα που σας ε, περιμένει ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προκλήσεις είναι πολλές. αλλά ευτυχώς για όλους μας, σε ένα μήνα από τώρα ένας ε, πολύ ικανός άνθρωπος ε, θα βρίσκεται ε, στο τιμόνι της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής Βοήθεια και της πολιτική προστασίας. Τον γνωρίζω καλά. και είμαι βέβαιος ότι με την εμπειρία του μπορεί να πετύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας, για την αφοσίωσή σας, για τη δέσμευσή σας ε, στο ε, ηθικό και ανθρωπιστικό μας πλαίσιο και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω, εφόσον μου το επιτρέψετε, ε, τις προσπάθειές μου στον τομέα αυτών. Ανά πάσα στιγμή θα είμαι στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων, για συζήτηση, για ανταλλαγή απόψεων. ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει όχι μόνο ο μεγαλύτερος χωρικός ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο, αλλά για να διατηρήσουμε και το ηθικό μας πλαίσιο, τις αρχές μας πάνω στην ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σας. Και φυσικά βλέπουμε ότι οι προσπάθειές σας ε, ε, απέναντι στον ιό έμπολα, τα συστήματα εκπαίδευσης σε ε, κρίσιμες καταστάσεις, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Και εγώ Σουηδός είμαι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που λάβαμε βοήθεια το 2018. Νομίζω ότι πάντα θα είσαστε ευπρόσδεκτος στη Σουηδία και πάντα θα είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών. Αναφερθήκατε και στη συνάντηση Ούγκα και είναι εξαιρετικό όχι μόνο ότι βλέπουμε την, την Ευρώπη να κατέχει ηγετική θέση, αλλά βλέπουμε και την ανάγκη η Ευρώπη να κατέχει ηγετική θέση στην ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Επίτροπε, δύο επιλογές έχετε. Ή θα θεωρήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόβλημα ή θα επιλέξετε να ε, συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική σας ε, επιλογή ήταν απόλυτα σαφής. Ε, δίνω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στυλιανίδη, νομίζω ότι δεν θεωρείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόβλημα. θα πρέπει να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, διότι περάσαμε δύσκολους καιρούς, γνωρίζουμε όμως και το τι πετύχαμε. Όπως ήδη ακούσαμε από σας, είχατε πάρα πολλή δουλειά τα τελευταία πέντε χρόνια και έπρεπε να αγωνιστείτε απέναντι στο κοινοβούλιο, απέναντι σε εμά, σε άλλους. Ελπίζω μόνο ο ε, διάδοχός να σας μοιάσει. Είχε καθυστερήσει το αεροπλάνο μου. Η πρώτη λέξη λοιπόν που άκουσα μπαίνοντας στην αίθουσα ήταν η εκπαίδευση από σας. και είμαι βέβαιος ότι θα διατηρήσουμε εδώ τα επιτέγματά σας. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η εκπαίδευση, η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, διότι τελειώς δεν υπάρχει βάση ούτε για αλλαγή ούτε για τίποτα. Το 2018 60 εκατομμύρια ε, παιδιών ε, δεν πήγαιναν ε, δημοτικό σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO. Είναι τραγικά τα νούμερα. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες. Αναφερθήκατε στην σημασία των πρώτων βοηθειών. Είναι και θέμα αξιοπιστίας. Ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Ε, είμαστε αδύναμοι, μερικές φορές έχουμε άδικο, ε, καταπολεμούμε ένα τον άλλον, αλλά υπάρχουν κάποια γενικά θέματα και όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να αναλάβουμε το ρόλο μας. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για μας, αλλά και για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πάντως, νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή βάση για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Νόισερ από το S&D. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Στην αρχή αναφέρατε τρία σημαντικά θέματα. Ξεκινήσατε από τον ιό έμπολα. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Δεν ε, λειτουργούσε τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ε, θερινές διακοπές ε, και δεν είχε αναλάβει ακόμα καθήκοντα ο νέος επίτροπος. Αλλά ήδη από την αρχή δείξατε πόσο δραστήριος άνθρωπος είσαστε. Η επίσκεψή σας στις χώρες αυτές ήταν επικίνδυνη, ήταν όμως και ένα σημαντικό μήνυμα ελπίδας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο η παρουσία σας το ίδιο είδαμε λίγες εβδομάδες μετά, όταν επισκεφτήκαμε και εμείς μια αντιπροσωπεία της ΔΕΒΕ, δηλαδή τις χώρες αυτές. Είδαμε πόσο σημαντική ήταν η αύξηση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ε, τόσο σημαντικό πρόβλημα. Είχαμε ανθρώπους σε καταβλισμούς Κανείς όμως δεν σκέφτηκε ότι έτσι θα έχουμε μία χαμένη γενιά χωρίς εκπαίδευση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ότι το επισημάνατε και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός ο τρόπος διαχείρισης από την πλευρά σας διότι συχνά έπρεπε να συνδυάσετε τις διάφορες απόψεις και ήταν πολύ σημαντικό το ότι τελικά καταφέραμε να εργαστούμε ως οικογένεια. Από διάφορα πολιτικά κόμματα ε, εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε σαν οικογένεια για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα σημαντικά για το μέλλον είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, διότι βλέπουμε όλο και περισσότερες κρίσεις. Ένα πρόβλημα όμως είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα διότι κοιτάνε τις κρίσεις ε, στην άμεση γειτονία τους και δεν, βλέπουν, βλέπουν τις κρίσεις ε, πιο μακριά. Τον Αμαζόνιο, τη Φουκουσίμα, το Μιανμάρ. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να ενεργήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι να δούμε απλά τι γίνεται έξω από την πόρτα μας, το οποίο είναι βέβαια σημαντικό, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και τις κρίσεις σε όλον τον κόσμο. Άλλωστε, είναι, θέμα των ευρωπαϊκών, είναι μέρος των ευρωπαϊκών αξιών το να δίνουμε ελπίδα. Νομίζω ότι ο διάδοχός σας θα πρέπει να μας πείσει θα πρέπει να εργαστεί σκληρά, να είναι αφοσιωμένος στο έργο αυτό. Εσείς μας δείξατε πώς μπορεί να ε, πετύχει πολλά ένας ε, επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση από τον κύριο αυτό. Από την κυρία Σιλβάνα Γκονσάλες από το S&D. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την εμπειρία που μας ε, ε, αναφέρατε. Εγώ ε, είμαι καινούρια στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό πραγματικά σας άκουσα με πολύ προσοχή και σας ευχαριστώ ε, για τα όσα μας είπατε. Ε, αναφερθήκατε και στην κλιματική αλλαγή, αναφερθήκατε στους ε, υποχρεωτικά εκτοπισμένους κλπ. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί δεν είναι μια κρίση πραγματικά, ε, είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει με πάγιο και συστηματικό τρόπο να αντιμετωπιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς πολλά εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν, να μετακινηθούν υποχρεωτικά τα επόμενα 50 χρόνια μάλιστα θα είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι αυτοί. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στην επόμενη θητεία και τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να βοηθήσει με συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης αναφερθήκατε στο Ρεσκυγιού Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια πολύ καλή πρακτική ε, της ε, Κομισιόν. Αλλά πώς πιστεύετε ότι μπορεί κανείς ή μπορεί ακόμα και το ίδιο το πρόγραμμα αυτό ε, να προχωρήσει απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά δεν έχουμε και νομική προστασία αυτών των ανθρώπων. Πώς νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο και μετά να ακούσουμε τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Σας παρακαλώ οι ερωτήσει να είναι πιο συντομέ όπω έκανε η κυρία Γκοντζάλας και για να μπορέσει και ο Επίτροπος να, κάνει τις, να δώσει τι απαντήσει του με σύντομο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια, για τη δουλειά που έκανα, όπως σας είπα. Ήταν μια κοινή προσπάθεια, κοινό το επίτευγμα όλα αυτά που κάναμε από την κρίση του έμπολα, ε, την ε, εκπαίδευση, τη u και πολλά άλλα και συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό μου φίλο. ότι συμπεριφερθήκαμε ως οικογένεια. Και αυτό ήταν το πιο βασικό στοιχείο για όλους μας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε και με τις υποχρεώσεις μας, αλλά και να έρθουμε στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Να ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Γκονσάλας για την αλλαγή του κλίματος. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα στην ΟΚΑ Ήταν πολύ ιδιαίτερη η συνάθρηση που είχαμε για την αλλαγή του κλίματος, αλλά ειλικρινά, γιατί πάντα είμαι ειλικρινής, στην οικογένεια αυτή τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής ήταν πραγματικά πιο χαμηλά από αυτά που αναμέναμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος και πιστεύω ακράδαντα ότι καταρχάς θα πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το στόχο αυτό, ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις μας με τους φίλους μας στην Ουάσιγκτον. Από πολιτικής άποψης, στη χώρα μου, ξέρετε, πάντα ήμουν υπέρ των υπερατλαντικών συμμαχιών. Αυτή είναι η πολιτική μου πεποίθηση. Και πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα της αλλαγής του κλίματος είναι πραγματικά αδύνατον. Δεν είναι εφικτό να πετύχουμε κρίσιμα αποτελέσματα χωρίς αυτή την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Συμμαχία. Άρα θα πρέπει να επιμείνουμε θα πρέπει να επιμείνουμε για να πείσουμε την κυβέρνηση Τραμπ σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα εφαρμογής της συνθήκης των Παρισιών. Όλα αυτά συνάδουν με τους στόχους μας και γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε, γιατί απλά ακολουθούμε τις επιστημονικές ε, τα επιστημονικά επιτεύγματα, τις επιστημονικές ε, γνώσεις, τα επιστημονικά στοιχεία. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να επιμένουμε για να μπορέσουμε να πείσουμε την Ουάσιγκτον για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την Συμφωνία του Παρισιού. Στην ε, συναντήσεις μου στην Ουάσιγκτον με τους ομολόγους μας, Είχα πολλές συναντήσει. συναντήσεις, συνδεθήκαμε πολλά άτομα που έχουν την ίδια ανησυχία. Όπως όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του κλίματος. Άρα, έχουμε πολλούς συμμάχους στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Κατά δεύτερον, πρέπει να ξεκινήσουμε, θεωρώ, όχι μόνο στα θεσμικά όργανα, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν μια απολύτως ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών θεσμικών οργάνων, της κοινωνίας των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα αυτό. Και όλα αυτά για να δούμε πώς μπορούμε βήμα-βήμα να προχωρήσουμε από κοινού. Δεν είναι δυνατόν πρόφανως παντού να υπάρξουν άμεσες δράσεις και αυτό θα πρέπει να το αναμένουμε, να προετοιμαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ξεκινήσουμε αυτόν τον ειλικρινή διάλογο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Εκ παραλίλου, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή αυτή η ευθύνη, είναι παγκόσμια. θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να λάβουμε κρίσιμες αποφάσεις. Ακόμα και αυτή τη μέθοδο κινήτρου και αντικινήτρου. Και σε αυτή να προσφύγουμε για να πείσουμε πολλούς ε, ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο για το πρόβλημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τον ανθρωπιστικό τώρα κλάδο. Να σας πω ότι η εμπειρία μου στην Αφρική, ιδιαίτερος, τι μου δείχνει ότι θα δούμε πολλά άτομα τα οποία θα είναι πρόσφυγες, ε, εσωτερικά εκτοπισμένοι, λόγω της αλλαγής του κλίματος. Δεν χωράει αμφιβολία. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος στην Αφρική. ή Ιδάλλως η κατάσταση θα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Και θα είναι όλο και πιο περίπλοκο να βρίσκουμε λύσεις. Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα, να δούμε τη ρίζα του προβλήματος. Τελευταίο σχόλιο για την Αφρική, όχι μόνο λόγω της αλλαγής του κλίματος, αλλά και για άλλους λόγους, δημογραφική ε, έκρηξη, διαφθορά, έλλειψη κράτους δικαίου. Άρα είναι τελευταίο σχόλιο είναι ότι ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την ε, τεράστια πρόκληση της Αφρικής, να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την Αφρική. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Η Αφρική για μένα δεν είναι μόνο μια ήπειρος, θεωρώ, προβλημάτων και προκλήσεων. Έχει και τεράστιο δυναμικό θα πρέπει να δούμε λοιπόν μια πραγματική εταιρική σχέση με την Αφρική, μια πραγματική συνεργασία πέρα από τη φιλανθρωπική προσέγγιση. Και φυσικά πέρα και από τα μετααπικιοκρατικά συμπλέγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και να συνεχίσουμε με ε, περαιτέρω ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Τέσσερις ερωτήσεις θα ακούμε κάθε φορά αν συμφωνείτε και μετά θα απαντάει ο Επίτροπος. Το μόνο το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φύγω στις 4.45 ε, γιατί πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Τέλεια, λέει ο Πρόεδρος. Να κάνουμε λοιπόν ε, κάποιες ε, γρήγορες ερωτήσεις. Έχουμε τέσσερις ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι οι πολιτικές ομάδες με έχουν μιλήσει. Να πάρει το λόγο η από τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ε, δέσμευσή σας, τη στράτευσή σας, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση, γιατί αυτό πραγματικά το συμμερίζομαι. Συμμερίζομαι αυτή τη θετική αιμονή όσον αφορά δε τις χώρες της Αφρικής. Είπατε ότι επισκεφθήκατε 55 χώρες, όχι μονάχα στην Αφρική και άλλες χώρες ε, και βοηθήσατε έτσι ώστε να αυξηθεί η βοήθεια για την εκπαίδευση ε, και ότι δώσατε δυνατότητα σε 5 εκατομμύρια νέους να εκπαιδευτούν. Ερώτηση. Διαπιστώσατε, αναφέρομαι κυρίως στις χώρες Σαχέλ, στις χώρες αυτές ε, διαπιστώσατε να υπάρχει η εκπαίδευση, η υποχρεωτική εκπαίδευση ε, υπάρχει λοιπόν υποχρέωση ε, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο γιατί εάν δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση ε, είναι δύσκολο να αυξηθεί ο ρυθμός των νέων που πηγαίνουν στο σχολείο. Εργαστήκατε, εργαστήκατε καθόλου για το θέμα αυτό. Γνωρίζετε λίγο τι γίνεται σε άλλες χώρες, όχι μόνο στις χώρες δηλαδή όπως το Ιράκ και το Ιράν που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένη κρίση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλτα Ιντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ανθρωπιστική βοήθεια και ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, θεμάτων όπως η υγεία ή η εκπαίδευση στα πλαίσια αυτά. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω ε, σε κάτι που αναφέρεται στο προγραμματικό σχέδιο της Φιλανδικής Προεδρίας και προκύπτει εκ νέου στην ε, Νιγηρία. Δηλαδή η συμφιλίωση ανάμεσα ή συντονισμός ανάμεσα ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιτρομοκρατική ε, δράση. Στην Νιγηρία είχαμε συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά απαγόρευση ε, των, της χρηματοδότησης συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα επίσης αντιτρομοκρατικά, ενώ διαπιστώνουμε ότι πάρα πολύ συχνά έχουμε την διάβρωση των μη κυβερνητικών ή ανθρωπιστικών οργανώσεων οργανώσεων από τρομοκράτες. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συστηματικά περνάει μπροστά από, από την ασφάλεια. Ε, βλέπουμε ότι και στην Συρία είχαμε παρόμοιες καταστάσεις όπου ε, βοήθεια ανθρωπιστική τελικά έφτανε ε, παράνομα στα χέρια των τρομοκρατών. Στο έγγραφο αξιολόγησης η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με τοπικούς εταίρου. Αλλά πώς διασφαλίζεται, εξασφαλίζεται η αξιοπιστία αυτών των τοπικών εταίρων όταν ξέρουμε ότι στους πολίτες των χωρών αυτών ε, τα τρομοκρατικά κινήματα είναι πολύ έντονα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις ε, πολύ σημαντικές παρατηρήσεις ε, που κάνατε. Ε, ε βεβαίως η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κατεξοχήν μικρής διάρκειας με την έννοια ότι είναι βραχυπρόθεσμη η αντιμετώπιση από την άλλη μεριά και εσείς αναφερθήκατε στην εκπαίδευση, στην δημιουργία υποδομών, την δυνατότητα να δοθούν ευκαιρίες ζωής σε πρόσφυγες δεύτερης γενιάς, σε ανθρώπους που θα εκτοπιστούν ή έχουν εκτοπιστεί ήδη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τι θα προτείνετε, τι θα συμβουλεύσετε ε, τον ε, διάδοχό σας, ε, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους κρίσεις, μήπως θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός του μακροπρόθεσμου με το βραχυπρόθεσμο και μια καινούρια αντιμετώπιση και των οικονομικών υποχρεώσεων. Ευχαριστώ κύριο Σταραμπέλα. Ε, ε, ε, εγώ θα ρωτήσω κάτι απλό ε, κύριε Επίτροπε. Εγώ βεβαίως ε, στην Επιτροπή ΑΣΕΑΝ ε, ταξίδεψα μαζί σας. Πήγαμε στην Τζακάρτα, πήγαμε σε, εκεί μετά από, από έναν σεισμό έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες κατασκευές με αντισυσμικά, αντισυσμικές πρωτεσίλες κλπ. Υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα μέσα στη δράση και την ε, επικοινωνία. Καλύτερα είναι δράση χωρίς επικοινωνία. Από την άλλη μεριά όμως, ε, μήπως υπάρχει και ένα έλλειμμα επικοινωνίας, δηλαδή μήπως υπάρχει και ένα έλλειμμα ορατότητας κάθε φορά που κάτι συμβαίνει ε, ε βλέπουμε τους Αμερικάνους ε, που κάνουν ολόκληρη ιστορία γιατί πετάνε μερικά αεροπλάνα τα οποία ρίχνουν κάποια κυβότια κτλ. Με βοήθεια. Ε, ε, είπατε ότι έχουν γίνει άμεσες παρεμβάσεις μέσω αυτών των νέων συστημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ευέλικτες, είναι άμεσες, είναι άμεσα αποτελεσματικές. Μήπως όμως πρέπει να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο την ορατότητά μας. Δεν λέω να το κάνουμε κάνουμε για λόγους, ε, πώς να σας το πω, publicity. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ε, θέλουμε να δούμε, ε, να βοηθήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους που, είναι, που έχουν αντιμετωπίσει καταστροφές, που είναι θύματα καταστροφών. Ευχαριστώ. Άλλη μία ερώτηση από, από την κυρία Σαμπό. Ευχαριστώ πολύ μία ερώτηση η οποία αφορά και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων αλλά και την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων. Λέω λοιπόν ότι μια ανθρωπιστική κρίση που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή όπως ας πούμε ε, η καταστροφή η ολιοσχερής ε, ενός νησιού το είδαμε στην νήσο του Σαν πριν από λίγο καιρό μετά από το πέρασμα ενός καταστροφικού ε, τυφώνα. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να υλοποιούμε τη Συμφωνία των Παρισίων με ταυτόχρονη ανθρωπιστική βοήθεια. Πριν από ένα χρόνο είχα τη δυνατότητα να πάω στην ολοσχερός καταστραφήσα νήσο του Σέμαρτα ε, και εκεί ε, δόθηκαν χρήματα ε, για την ανακατασκευή, αλλά δυστυχώς οι νέες κατασκευές ήταν ακριβώς όπως οι προηγούμενες. Μήπως πρέπει κάπως να μάθουμε από τα διδάγματα τέτοιων καταστροφών έτσι ώστε να αλλάξουμε μοντέλο και αυτά τα διαφορετικά μοντέλα να ληφθούν υπόψη. Εγώ είχα ε, υποβάλει τον προηγούμενο Ιούλιο ε, μία έκθεση κατά πρόταση κατά την έννοια αυτή. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει. Και να κλείσει και τη συζήτηση και ελπίζω έτσι να προλάβουμε στις 5 να είμαστε έτοιμοι. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Αγαπητέ συνάδελφε, σχετικά με το νέο τρόπο σκέψης για το κλίμα, για το περιβάλλον. Ειλικρινά, δεν είμαι εμπειρογνώμων. ούτε προσπαθώ να δείξω ότι είμαι εμπειρογνώμων. Τα τελευταία πέντε χρόνια κατέβαλα προσπάθειες για να συγκεντρώσω ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων για το θέμα αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω πραγματικά ότι η Συμφωνία του Παρισιού ήταν σημαντικό επίτευγμα ιδιαίτερα της Ευρώπης διότι πιθανότατα γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι στο Παρίσι καταφέραμε να σπρώξουμε όλον τον κόσμο για να, πετύχει, για να δεχτεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για την αλλαγή του κλίματος. για τη δική σας προσέγγιση μπορώ να πω το εξής, ότι μέσα από το Rescue μέσα από τη νέα δομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όχι μόνο έχουμε περισσότερα αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά εστιάζουμε εξίσου στην πρόληψη και την ετοιμότητα. Και για μένα, αυτός ο τρόπος σκέψης, όπως ακριβώς είπατε, είναι ο πιο σημαντικός. Πρέπει να εστιάσουμε και στην πρόληψη και την ετοιμότητα για να αλλάξουμε πολλά πράγματα στις κοινωνίες μας και στην αντιμετώπιση μας απέναντι στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, δασικές πυρκαγιές. Σε πολλές μεσογειακές χώρες χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά ε, στους πρώτους που ε, επεμβαίνουν, ε, στους εθελοντές, ιδιαίτερα στις υπαίθριες περιοχές, στις αγροτικές περιοχές. Από την άλλη, πρέπει να βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε ε, τα δάση με αντιπυρικές ζώνες, με διαδρόμους για να μπορούν να περάσουν ε, τα πυροσβεστικά οχήματα. Μιλάω για πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά θέματα. Επίσης, ε, για, ε, για σεισμούς. Κάθε τέτοιο γεγονός χρειάζεται νέα προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη, διότι όπως είπαμε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αλλαγή του κλίματο, πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Πρέπει να συνδυάσουμε αυτό με νέα εργαλεία για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο κάθε φυσικής καταστροφής. Χωρίς όμως πρόληψη και ετοιμότητα, Κανένα μέσο, κανένα αεροπλάνο, ελικόπτερο δεν αξίζει τίποτα. απέναντι σε μια φυσική καταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με την πρόληψη και την ετοιμότητα και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές κλπ. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι ένα στρατηγικό σχέδιο Χρειαζόμαστε όμως πρόληψη και ετοιμότητα και χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα μέσα για να σώσουμε ζωές και να περιορίσουμε ε, τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Εγώ πιστεύω σε μια τέτοια ολιστική προσέγγιση και η Ευρώπη, ναι, παραμένει πρωτοπόρος σε όλα αυτά. Ένα πράγμα χρειάζεται μόνο να σας πω ότι ακόμα και οι Πολιτείες επανειλημμένα Μα έχουν ζητήσει το εξαιρετικό σύστημα χαρτογράφησης Κοπέρνικους για να αντιμετωπίσουν τι δασικέ πυρκαγιέ στην ε, Καλιφόρνια, ε, τις πλημμύρε ε, στο Τέξας κλπ. Έχουμε λοιπόν σημαντικά εργαλεία στο διάθεσή μας που μπορούμε να προσφέρουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Κυρία Ταραμπέλα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και ένα από τα προβλήματά μου ήταν αυτό που είπατε. Δεν κατάφερα να έχω μεγαλύτερο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια. Δαπάνησα πολύ χρόνο, πολύ προσπάθεια. Υπάρχει όμως μια παράδοση κάποιοι από τους εταίρους μας στην ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα να είμαι και σαφής. Πιστεύουν ότι όταν θέλουμε να αυξήσουμε την ορατότητά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσουμε την ιδιωτερότητά μας και την αμεροληψία μας. Εγώ διαφωνώ τελείως. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειάζεται να είμαστε πιο ορατοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για πολλούς λόγους και όχι μόνο εντός Ευρώπης αλλά και εκτός διότι είμαστε οι μόνοι που επιμένουμε πάνω σε ένα ε, πλαίσιο παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα πλαίσιο αρχών. Μια συμβουλή μου λοιπόν προς τον διάδοχό μου είναι να αυξήσει την ορατότητά μας ε, και σας παρακαλώ να τον βοηθήσετε σε αυτό. Αγαπητέ φίλε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπατε τα πάντα. Αναφέρατε την πιο σημαντική λέξη, την σύνδεση ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή βοήθεια, νέξους. Ε, είναι μια μαγική λέξη στις συζητήσεις μας και πρέπει να τη νιώσουμε. Διότι σε μεγάλο βαθμό παραμένει και από νόημα. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση σε περιπτώσεις κρίσεων είναι ο ορισμός αυτής της σχέσης ανάμεσα στην ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτή ήταν η προσέγγιση μου ήδη από την αρχή της ε, θητείας μου. Το Rescue και όλα αυτά τα θέματα. Αυτός, αυτή είναι η σημαντική πρόκληση για όλη την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για όλους όσους διαμορφώνουν την πολιτική. Θα πρέπει να νιώσουν ε, το nexus, ε, το, τη σύνδεση αυτή. Πρέπει να καταργήσουμε ε, τα σιλό, τους απομονωμένους τομείς. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοια, τέτοιους απομονωμένους τομείς, ε, δεν επιτρέπεται να έχουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχω καταβάλει πολλές προσπάθειες τα τελευταία πέντε χρόνια σε συνεργασία με πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με τον Γενικό Διευθυντή ε, των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες, ε, γνωρίζει τα θέματα αυτά, διότι ήταν διευθυντής ε, του UNHCR. Καλό και σας, σας παρακαλώ, ασκήστε πίεση για να βρεθούν πρακτικές λύσεις, ώστε να έχουμε στην πράξη σύνδεση ανάμεσα στους τομείς αυτούς. σχετικά με τη ζώνη Σαχέλ και ε, της ε, κρίσης εκεί. Έχω επισκεφτεί επανειλημμένα χώρες ε, της περιοχές Σαχέλ, το Νίγηρα, το Τσάντ, το Μάλι και είδα τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους ιδιαίτερα για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Γνωρίζετε ότι ο βασικός πυλώνας για οποιαδήποτε βελτίωση ε, του βιωτικού επίπεδου στη περιοχή αυτή είναι τα κορίτσια και οι γυναίκες. Ξεκινήσαμε, αυξήσαμε ε, τον προϋπολογισμό ε, για τις κρίσεις, για τις οξύες κρίσεις, αλλά τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό για τις γυναίκες, για την εκπαίδευση των κοριτσιών και μέσα από αυτήν την προσέγγιση να μειώσουμε τους ε, ε, γάμους σε μικρή ηλικία και τους ε, καταναγκαστικούς γάμους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα στα χωριά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ θερμά. Πρέπει να βρούμε εταίρους ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις ε, και άλλους φορείς στην Ιγυρία κλπ. Πιθανότατα να μην το ξέρετε, αλλά στο κύριο Νούγκα, μαζί με το Βέλγιο, είχαμε οργανώσει μια εξαιρετική εκδήλωση για την αντιτρομοκρατία, την ανθρωπιστική βοήθεια και όλες τις πτυχές του θέματος αυτού. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά και όλες τις ομιλίες, διότι είχαμε εξαιρετικούς ομιλητές που γνωρίζουν τα θέματα αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Όλοι όμως ε, συμφωνούσαν στο εξής. Άσχετα από τους κινδύνους συμμετοχής τρομοκρατικών οργανώσεων στην ανθρωπιστική μας βοήθεια. Οι στόχοι μας ξεπερνούν αυτό το μικρό και συχνά άσχετο με το θέμα μας ε, θέμα. Πρέπει να αναλάβουμε τον κίνδυνο. Συχνά πρέπει να είμαστε σε, επαφές, ε, σε επαφή με τις αρχές για να περιορίσουμε το πρόβλημα αυτό αλλά δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιούμε αυτό ως δικαιολογία για να περιορίζουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Επιτρέψτε μου να πω μόνο δύο λόγια να κάνω μια μικρή σύνοψη, αν μου επιτρέπετε. We had a challenging task. Ήταν απαιτητική η δουλειά που είχαμε να κάνουμε τα πέντε χρόνια αυτά. Για να συνοψίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε πάρα πολλούς ε, εταίρους και χιλιάδες ε, εμπειρογνώμονες και συναδέλφους. Αν μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τους συναδέλφους μου στην ΕΚΟ. Δύο εξ αυτών είναι και εδώ, παρόντες σήμερα στην αίθουσα. Δεν θέλω να είμαι μεριληπτικός για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά μπορώ να πω, το ξέρουν και οι φίλοι από τη γραμματεία, ότι στις υπηρεσίες μας, στην ΕΚΟ, ιδιαίτερος και στο ERCC, στο κέντρο κατεπίγουσας ανάγκης, είμαστε πολύ τυχεροί λόγω των γνώσεων, των ικανοτήτων και των προσπαθειών που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί μου φίλοι. Just to say few... Και να πω λοιπόν δύο λόγια για κάποιες πρωτοβουλίες μέχρι στο τέλος της θητείας αυτής. Στα τέλη Οκτωβρίου με την ύπατη εκπρόσωπο Φεντρίκα Μοτογίνη. Εδώ στις Βρυξέλλες θα οργανώσουμε μία συνεδρίαση αλληλεγγύης για τη Βενεζουέλα με την UNHCR και την την IOM. Θα είναι και η τελευταία εκδήλωσή μας. Για το 2019. Τον Οκτώβριο λοιπόν. Τέλη Οκτωβρίου. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο τομείς, ε, κάποιους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επιμείνετε για να βρείτε λύσεις. Ενδεχομένως να επισκεφτείτε και τις περιοχές αυτές για να μπορέσετε να αξιολογήσετε την ε, κατάσταση. Η Εμένη, Αφγανιστάν, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, Ουκρανία. Είναι μεγάλος ο κατάλογος ε, των συγκρούσεων. Και εκεί βλέπουμε πραγματικά ανθρώπινο πόνο πέρα από κάθε φαντασία. Είναι καλή ιδέα αυτή για την προβολή του έργου μας να παραστεί τόπου η Επιτροπή ΔΕΒΕ με ή χωρίς τον Επίτροπο να υπάρχει μια ομάδα. Αλλά εκ παραλλήλου θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει και κάποια αρχή αν θέλετε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Τα πολιτικά προβλήματα, ξέρετε, δεν μπορούν να επιληθούν με ανθρωπιστικές λύσεις και τα ανθρωπιστικά προβλήματα χρειάζονται πολιτικές λύσεις. Άρα, συνεχίζουμε το ανθρωπιστικό μας έργο σε κάθε περίπτωση, πέρα από κάθε αμφιβολία. Επιμένουμε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών, αλλά εκ παραλλήλου σε Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε και μία συνολική προσέγγιση από πολιτική άποψη σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ανάπτυξη χρειαζόμαστε αυτή τη δετή προσέγγιση. Είναι λοιπόν κρίσιμο αυτό για μας ως ε, πολιτικοί θύγνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτική προσέγγιση. Είναι άλλωστε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα για σήμερα και για αύριο. Η νέα Επιτροπή έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ανθρωπιστικών κρίσεων να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς θα έχετε μια βεβαρημένη ατζέντα στο μέλλον. Έχουμε προλιάνει όμως το έδαφος και γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Οι λαοί μας, οι πολίτες μας δεν θέλουν άλλο μπλα θέλουν συγκεκριμένες δράσεις, ιδιαιτέρως στο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, καλύτερα να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αγαπητοί φίλοι, πριν από πέντε χρόνια με εμπιστευτήκατε για να γίνω το πρόσωπο της ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλο τον κόσμο. Ήταν η ύψιστη τιμή στη ζωή μου. πέρα των πολιτικών ευθυνών. Η θέση αυτή ήταν πραγματικά ύψιστη στην τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι που σταθήκατε στο πλευρό μου σε όλη αυτή την ε, μεγάλη και πολύπλοκη διαδρομή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας και το δηλώνω αυτό ενώπιον της Επιτροπής ΔΕΒΕ ότι ήσασταν πραγματικά πολύ κοντά στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Commissioner, uh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα βέβαια εξ ονόματος της Επιτροπής μας ε, να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας ε, για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ξέρουμε ότι Είστε πολύ θεσμευμένος με τα θέματα αυτά, γι' αυτό φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι θα σας συναντήσουν όσον ούπο. Ε, καλή συνέχεια λοιπόν. Ναι, όποτε θέλετε, εγώ μπορώ να είμαι στη διάθεσή σας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε λοιπόν και τώρα θα μετακινηθούμε στην κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ και ε, την Ντρουά. Ε, και θα συζητήσουμε για την υποψηφιότητα των βραβείων Ζαχάροφ. Παρακαλώ, θα μετακινηθούμε. Τα λέμε σε λίγο.